Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε την μερίσια διάταξη. Θα συνεχίσουμε το σημείο 14, που είναι η παρουσίαση του συστήματος της Εστονίας για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Πρέπει να σας πω ότι Έχω ήδη μεταβεί δύο φορές στην Εστονία επί Εστονικής Προεδρίας. Την πρώτη φορά που πήγα ήταν το άτυπο ε, Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εστερικών Υποθέσεων, όπου μας ε, παρουσιάστηκε αυτό το σύστημα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην Εστονία και πραγματικά με κατέπληξε η παρουσίαση αυτή. Επίσης, μια δεύτερη παρουσίαση ήταν η ψηφιοποίηση γενικά της κρατικής διοίκησης στην Εστονία, που και αυτό με κατέπληξε. Δεύτερη φορά έμεινα έκπληκτος και θεώρησα ότι θα είναι καλή ιδέα να μάθετε κι εσείς τι κάνουν στην Εστονία και να εκπλαγείτε κι εσείς. Καλωσορίζω λοιπόν με μεγάλη χαρά την κυρία Κέτλεν Κατάη, που είναι η επικεφαλής ε, του Κέντρου Εθνών Σχέσεων μιας ε, οργάνωσης ε, που πληροφορικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα της δώσω της κυρίας κατευθείαν το λόγο. Όπως πολύ σωστά σας είπε ο Πρόεδρος, λέγομαι Κάτλιν Κέτεϊ και είμαι υπεύθυνη διεθνών σχέσεων σε ε, ένα κρατικό φορέα πληροφορικής που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Εστονίας. Μου ζητήθηκε σήμερα, μετά την συνεδρίαση του άτυπου συμβουλίου που σας ανέφερε ο κύριος Σφόποντα, να σας παρουσιάσω μια μελέτη περιπτώσεων που είχα παρουσιάσει τον Ιούλιο στην Εστονία αλλά καταρχάς να πω ότι η υπηρεσία μας παρέχει υπηρεσίες πληροφορικές, δηλαδή ασχολούμαστε με ό,τι έχει να κάνει με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και όταν μας στήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Εστονίας να παρουσιάσουμε ένα μελλοντικό ε, σενάριο ενδεχομένω ε, τον Ιούλιο, γενικότερα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ένα υποθετικό σενάριο, εγώ άρχισα να βλέπω τα πράγματα από την πλευρά των πολιτών. Διότι τελικά αυτή είναι που είναι στο επίκεντρο. Και οι καταναλωτέ, ή μάλλον συγγνώμη, και οι επιχειρηματίε που θα είναι στο επίκεντρο θα χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Και καλό να κάνουμε τη ζωή του όσο το δυνατόν πιο άνετη και ασφαλή. Τον Ιούλιο, λοιπόν, κατέληξε μια αποθετική μελέτη περιπτώσεων. Πάντα από το πρίσμα των πολιτών τη Ένωση για το πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα ευρύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Διότι ο στόχος από την πλευρά των πολιτών πάντα είναι να μπορούν να επικοινωνούν με οποιοδήποτε φορέα και θεσμό, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κρατικό, με έναν γρήγορο, ασφαλή και ιδεατά ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς χαρτί. Αυτό είναι πιο γρήγορο και πιο οικονομικό και για τον πολίτη και για το κράτος. Αρχικά λοιπόν αλλάζουν διαφάνειες. I first to a... Ο στόχος που φαντάστηκα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι στόχο θα έπρεπε να έχουμε, γιατί αν δεν έχουμε θα χαθούμε εύκολα. Και θα μας απογοητεύσουν τα μικρά εμπόδια και θα χάσουμε τη γενική εικόνα. Άρα ο στόχος που σκέφτηκα είναι να έχουμε ανοιχτή ψηφιακή δικαιοσύνη για όλους. Και όταν λέω ανοιχτή δικαιοσύνη, όχι προσβάσιμη, αλλά οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να δει κάποιες πληροφορίες, να μπορεί να βλέπει τα ίδια δεδομένα την ίδια χρονική στιγμή. Κατά την άποψή μα, στην Εστονία αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ολοκληρωμένε ηλεκτρονικέ υπηρεσίε που θα δίνουν στον πολίτη τη δυνατότητα να επικοινωνεί με το κράτο, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ηλεκτρονικά χωρίς ε, έντυπα έγγραφα. Ας φανταστούμε κάτι άλλο σε σενάριο. Συγκροτείται μια εταιρεία από έναν Ευρωπαϊκό πολίτη. Κατά το αισθονικό δίκαιο στην προηγούμενη υπόθεση αυτή. Θα μπορούσε αυτό να γίνει με σύνδεση σε ένα πόρταλ, σε μία πύλη, ώστε να μπορεί κανείς ηλεκτρονικά εντελώς να συστήσει την εταιρεία με την εθνική ταυτότητα. Συνδέεται σε αυτό το σύστημα. Και αφού συνδεθεί στο σύστημα, το σύστημα ζητά από το μελλοντικό επιχειρηματία τι είδος εταιρεία θέλει να ιδρύσει. Εταιρεία περισμένης ευθύνης, ιδιωτική αυτή διαλέξαμε εδώ έτσι, για λόγους ευκολίας. Τέσσερα βήματα μετά ε, είναι η διαδικασία που καλείται να φέρει σε πέρας αυτός ο επιχειρηματία. Πρώτον, να συμπληρώσει τα στοιχεία, ε, ονομασία, καταστατικό ε, οικονομικό έτος, οικονομική χρήση και για να μπορέσει να είναι διαθέσιμη αυτή η πύλη σε διάφορες γλώσσες. Ο μελλοντικό επιχειρηματίας μπορεί να καταναλώνει εντό αγωγικών και να χρησιμοποιεί αυτή την πύλη στη γλώσσα του. Και στην προκειμένη περίπτωση τα ίδια δεδομένα να τα βλέπει και στην επίσημη γλώσσα του κράτους. Αυτό είναι πιο απλό για την χώρα αλλά και για τον πολίτη που είναι και ο τελικός στόχος. Αφού λοιπόν γίνει αυτό των δεδομένων, πρώτο βήμα, το δεύτερο, δεύτερο είναι το σύστημα ε, παράγει ε, ένα cover letter προς το πρόσωπο που θέλει να συγκροτήσει ε, το νομικό αυτό πρόσωπο. Τα μεταδεδομένα τα έχει βάλει ήδη ο πολίτης από πριν στο σύστημα και τα άλλα τα αναλαμβάνει το σύστημα. Ο πολίτης επίσης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί με την ηλεκτρονική υπογραφή να συστήσει την εταιρεία. Πάντα μέσω τη εθνική ε, ταυτότητα μπορεί να γίνει αυτό, βάζοντα το δεύτερο κωδικό PIN. Νομικά δεσμευτικό αυτό και το σύστημα περνάει αυτόματα στο σύστημα 3, που είναι η καταβολή του τέλους, του κρατικού τέλους. Δηλαδή να μην λαμβάνονται αναφορές που θα λένε ότι δεν έχει πληρωθεί αυτό το τέλος. Και έπειτα κάθεται και περιμένει την επιβεβαίωση της κυβέρνησης επιχειρηματίας και ελπίζει να πάρει θετική απάντηση. Σποθέσουμε ότι αυτή η διαδικασία κρατάει καμιά δυο ώρες το πολύ. Για λίγες ελάχιστες μέρες. Και μετά ιδρύεται η εταιρεία. Ας πούμε ότι είναι στην κινητή τηλεφωνία η επιχείρηση αυτή και τα πάει καλά στην αρχή. Όμως αυξάνονται οι δυσαρεστημένοι πελάτες και κάποια στιγμή από τους πολίτες, πολύ δυσαρεστημένος πελάτη που δεν μπορεί να καταλήξει σε μια αμοιβαία ε, συμφωνία, ε, μηνύει την ε, εταιρεία. Αλλά πρώτα θέλω να αυτοί οι συγκεκριμένοι πελάτες να πούν αν είναι οι πρώτοι ή υπήρξαν και άλλες υποθέσεις, υπήρξαν και άλλοι δυσαρεστημένοι. Πάνε λοιπόν στην πύλη αυτή του e-justice και ψάχνουν με το όνομα της εταιρεία για να δουν κατά πόσον υπάρχουν και άλλες δικαστικές υποθέσεις με αυτή την εταιρεία. Και βρίσκει μια λίστα που δείχνει ότι ορίστε υπήρξαν και κατά το παρελθόν δικαστικές υποθέσεις, διαφορές της εταιρεία με πολίτη Και αυτή είναι η σταγόνα που κάνει το ποτέρι, ξεχυλίζει για τον πολίτη και κάνει την προσφυγή στο δικαστήριο κατά της εταιρεία. Πρώτα τι κάνει, μπαίνει στο σύστημα, συνδέεται με την εθνική ταυτότητα και αρχίζει να υποβάλλει αυτό το κείμενο, παραδείγματος χάρη αστική ε, δίκη διαλέγει το έγγραφο, το δικόγραφο. Τι είδου υπόθεση και σε ποιο δικαστήριο θέλουν να συζητηθεί η υπόθεση, ανάλογα με το που βρίσκονται και οι ίδιοι που θα μπορούν να πάνε, να παραστούν. Και το σύστημα ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο. Μπαίνει ένα αρχικό ποσό για την προσφυγή Μπορεί κανείς να προσθέσει επίσης ε, άλλους ε, πέραν των δύο διαδίκων ενδεχομένως και άλλους που θα συμμετέχουν. Μετά αναρτάται αυτή η υπόθεση, το δικόγραφο, ενώ στο μέλλον θα μπορούσε το σύστημα να ρωτάει κι άλλα, να κάνει κι άλλες ερωτήσεις και με βάση τις απαντήσεις να παράγει αυτόματα το φάκελο της δικογραφίας. Μετά με internet banking καταβάλεις το τέλος και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η πύλη που δουλεύει στο υπόβαθρο. Το σύστημα πληροφοριών της πύλης δίνει έναν ενιαίο μοναδικό αριθμό στην υπόθεση, την στέλνει στο αρμόδιο δικαστήριο και κοινοποιεί στο τμήμα αυτό του δικαστήριου ότι έχετε μια νέα υπόθεση. Μέχρι στιγμής ούτε μία σελίδα χαρτί δεν χρειάστηκε. Το δικαστήριο βλέπει τα έγγραφα και επίσης το σύστημα βλέπετε εδώ ότι αυτό με το κίτρινο είναι ακριβώς η υπόθεση αυτού του δυσαρεστημένου πελάτη. Βλέπει λοιπόν το δικόγραφο το δικαστήριο, έχει την ίδια ημερομηνία, αλλά σε ένα άλλο, σε μια άλλη διαπαφή χρήστη, για να είναι στο δυνατόν πιο εύκολο να το διαχειριστεί και να το μελετήσει. Και αν θεωρηθεί ότι είναι βάσιμη η καταγγελία και με βάση και τις πληροφορίες εκδίδεται δικαστική εντολή, διαταγή να ξεκινήσει δηλαδή η δίκη και το σύστημα με βάση τα μεταδεδομένα συμπληρώνει τις πληροφορίες σε μεγάλο βαθμό και τι απομένει για τον κλητήρα, για τον ε, γραμματέα του Καστήλ, να βάλει ένα, ε, να συμπληρώσει δύο τετραγωνίδια που θα πάνε τα στοιχεία για τον ε, ενάγοντα και τον εναγόμενο. και τα άλλα τα αναλαμβάνει το σύστημα. Εγώ τώρα είμαι ο δυσαρεσμένος πελάτη και περιμένω κοινοποίηση από το δικαστήριο για να δω αν έχει ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Ξαναπάω σε αυτή τη διαπαφή και βλέπω ότι έχει έρθει ένα νέο έγγραφο, όπως βλέπετε με τον κλειστό φάκελο και στην οθόνη. Το ανοίγω το έγγραφο που σημαίνει ότι μου είχε επιδοθεί και ξεκινάει να τρέχει ημερομηνία, η προθεσμία από τότε. Επίσης, στο υπόβαθρο το σύστημα πληροφοριών σώζει τις ημερομηνίε. και προχωράει. Η υπόθεση φτάνει στο τελικό στάδιο ηλεκτρονικά διαβιβάζεται η τιμιγόρια του δικαστηρίου στα μέρη στην πύλη. Όπως είδαμε πριν έρχεται το πρώτο έγγραφο, έτσι φτάνει και η τιμιγόρια του δικαστηρίου. Φυσικά αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά σήμερα στην Εστονία δεν είναι science fiction, είναι πραγματικότητα. Το χρησιμοποιούμε σήμερα αυτό το σύστημα στη χώρα μας. Κατά κόρον. Και υπεύθυνη για την διατήρηση και την επεξεργασία αυτού του συστήματος είναι η δική μας υπηρεσία. Δεν ξέρω τελικά πόσο απέχουμε από το στόχο μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί σήμερα ήδη, ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά. Έχουμε το e codex τον ανταλλαγή δεδομένων. Έχουμε το e idis Άρα έχουμε ξεκινήσει να βάζουμε κάποια λιθαράκια για τον επιτεύξη του στόχου που ανέφερα στην αρχή της παρουσίασης. Επίσης, ως κρατικός φορέας στην Εσθονία φυσικά και μας ήταν πολύ πιο εύκολο να αναπτύξουμε αυτά τα συστήματα. Για τη σπονδυλική στήλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Εστονία παρέχεται και διατηρείται κεντρικά στην κυβέρνηση, από την κυβέρνηση. Ποια είναι αυτή η σπονδυλική στήλη, ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρώτον, η ηλεκτρονική ταυτότητα, το X-Road διάφοροι φορείς με λίγο κόστος και με αποτελεσματικό αποκεντρωμένο τρόπο μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων μητρών και συστημάτων πληροφοριών με ασφαλή αποκεντρωμένο τρόπο, όπως είπα. Επίσης, αν αυξάνονται οι πληροφορίες και τα μητρώα, πάλι μπορεί κανείς εύκολα να χάσει την γενική εικόνα. Δηλαδή να υπάρχουν δεκάδες ή χιλιάδες μητρώα που να συλλέγουν τι πληροφορίες. Η λοιπόν διάλεξε να υπάρχει ένας εθνικός κατάλογος ε, συστημάτων πληροφορικής ή μητρών με στόχο πρώτο. Κάθε νέο σύστημα πληροφορίας πρέπει να εγκριθεί, δηλαδή να πάρει το πράσινο φως να δημιουργηθεί όχι. Μπορεί να προκύπτει στοιχεία στο δημοτολόγιο και με το X-Road μπορεί εύκολα να ζητηθεί. Αλλά έχουμε αυτό το ρίχα, που είναι αυτό το εθνικό, εθνικό κατάλληλο, μπορεί να λέει δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα. Μετά, έχουμε αποκεντρωμένη διασύνδεση των συστημάτων. Για να δούμε ποιο μητρό έχει ποιο στοιχείο. Αυτός είναι ένας στόχος. Άλλος στόχος όμως. Αντί να ζητάμε τα ίδια δεδομένα ξανά και ξανά από τον πολίτη, στην Εστονία επιλέξαμε μια άλλη οδό. Να γίνει αυτόματα με το στρώμα αυτό της ανταλλαγής σε ηλεκτρονικά πληροφοριών αυτή η αίτηση. Επίσης και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων κρατικών φορέων είναι δωρεάν. Γιατί ο πολίτης είναι ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος των δεδομένων και όχι το κράτος η κυβέρνηση. Επίσης η Ιστονία έχει θέσει και κάποιους στόχους, όχι κανόνες, κάποιους ε, στόχους για το ψηφιακό θεματολόγιο. Έχω κάποιους από αυτούς στη διαφάνεια αυτή που νομίζω ότι σχετίζονται λίγο πολύ. Θέλουμε να υπάρχει διαλειτουργικότητα όχι μόνο εντός των συνόρων, αλλά και διασυνοριακά. Αυτό το στόχο φέτος το Μάρτιο ο Υπουργό ε, Οικονομικών Εστονία με τον Υπουργό Οικονομικών Φιλανδία υπέγραψε μια συμφωνία για να αρχίσουν να ανταλλάσσουν από το φθινόπωρο στοιχεία. Ελπίζουμε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να γίνει πραγματικότητα η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών. Προς αυτό εργαζόμαστε. Και για μας αλλά και για τον πολίτη το σημαντικό είναι να μην ε, μπίνουμε στην παρο... να μην ε, κολλήσουμε στην παροχημένη, ξεπερασμένη τεχνολογία. Φυσικά και μπορεί κανείς να βελτιώνει τα συστήματα. Αλλά αν μετά από 13 χρόνια την περίπτωση τη Εστονία, α πούμε, έχει παλιώσει το σύστημα, δεν μπορεί να το μπαλώνει και να το ξαναμπαλώνει. Αλλά καλύτερα να το ξεφορτωθεί στο παλιό σύστημα και να δημιουργήσει ένα τελείω διαφορετικό σύστημα, μια νέα αρχιτεκτονική, μια νέα τεχνολογία. Για να είναι ασφαλέ και αποτελεσματικό αυτό το σύστημα. Πολλά τα αστυνομικά σήμερα είναι ηλεκτρονικά μόνο διαθέσιμα. Όπως το κτηματολόγιο ή το μητρό εταιριών. Είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο που τον Ιούνιο φέτος υπέγραψε μια συνθήκη για να ανοίξει μια ψηφιακή πρεσβεία. Θα στηρίζει αυτά τα δεδομένα. Στο Λουξεμβούργο βεβαίως θα, γίνει, θα ανοίξει το, η πρώτη τέτοια πρεσβεία. Επίσης, οποιοδήποτε στον κόσμο μπορεί να γίνει πολίτης Εστονίας με το e-residency που έχουμε από το Δεκέμβριο του 2014. Παίρνει ηλεκτρονική ταυτότητα και μπορεί να έχει πρόσβαση στα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Two slides on our institution. Δύο διαφάνειες τώρα για το φορέα μας, για να καταλάβετε γιατί εμείς ε, αναλάβαμε παρουσιάσουμε αυτό το υποθετικό σενάριο. Με την αύξηση των συστημάτων πληροφοριών και στο νομικό τομέα, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών για να μπορεί να υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Εμείς είμαστε μια υπηρεσία πληροφορικής αλλά η μισή είναι νομική. Έχουν πάνω από 200 επαγγελματίε στην υπηρεσία μας. Και με αυτούς διατηρούμε πάνω από 70 συστήματα πληροφοριών πολύ σημαντικά για τον πολίτη και για το κράτος. Σας έδειξα ποια είναι τα σημαντικά από αυτά, τα πιο σημαντικά από αυτά και εδώ βλέπετε και μερικά ακόμη σημαντικά συστήματα πληροφόρων που κατά είναι ο πυρήνας της ανοιχτής δικαιοσύνης, ε, της ε, προσβάσιμης δικαιοσύνης στην Εστονία. Φυσικά και δεν ήταν εύκολο, είχαμε εμπόδια να αντιμετωπίσουμε, δώσαμε μάχες. Μπορεί να υπήρχαν ε, εμπόδια δημοσιονομικά, ανάλογα με τις επιθυμίες, τις διαφορετικές απόψεις κτλ. Αλλά η εμπειρία μας μας έχει διδάξει ότι αντί να εστιάζουμε στο τι δεν μπορούμε να πετύχουμε, καλύτερα είναι να εστιάζουμε στο τι μπορούμε, ποιες λύσεις μπορούμε να βρούμε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το ΡΙΚ, το κέντρο μας, μόνο, και για την Εστονία εν γέννη και θα ήθελα να ελπίζω και να πιστεύω γιατί όχι να μην ισχύσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Πράγματι, η ασθενεία είναι τόσο ψηφιακή που πρέπει να διασφαλίσω, να διαβεβαιώσω ότι η κυρία Κατά είναι εδώ η ίδια και δεν έχουμε μια εικονική παρουσία της. Λοιπόν, για να κατανοήσουμε πώς ε, λειτουργεί η Εστονία βάθος, ε, έχουμε δύο ερωτήσεις κατά νου. Καταρχήν, πώς είναι δυνατόν η Εστονία με κάθε σεβασμό δεν είναι μεταξύ των ε, πλούσιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τα έχει καταφέρει και μπορεί τα μέλη να αναρωτιούνται σχετικά με το θέμα της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων στο σύστημα. Από όσο γνωρίζω, η Εστονία έχει επιλέξει πολύ διαφορετική λύση από τον περιορισμό. Δίνει αντιθέτως πρόσβαση σε όλα τα άτομα στα προσωπικά τους δεδομένα. Και φυσικά και αυτός ε, ο κατάλογος ετοιμάτων είναι διαθέσιμος ε, και επιγραμμικά. Αλλά να μας εξηγήσετε γιατί η Εστονία. Δύσκολη ερώτηση. Ελπίζω ότι είναι χάρη στην οτροπία. Δηλαδή δεν είχαμε και πολλή επιλογή στην αρχή, παρά να είμαστε αποτελεσματικοί. Όπως σωστά είπατε, η Εστονία δεν είναι μεγάλη χώρα, ούτε από διεσυνοσιονομική, ούτε σκοπιά, ούτε από τη σκοπιά πληθυσμού. Με 1,3 εκατομμύρια πληθυσμό πρέπει να είμαστε αποτελεσματική και η Ιστονία προσπαθεί να έχει ως το δυνατόν μικρότερο δημόσιο τομέα. Βέβαια, αυτό ε, σημαίνει ότι για κάθε κυβέρνηση ήταν προτεραιότητα η ψηφιοποίηση για 50 χρόνια, συγγνώμη, για 15 χρόνια τώρα υπήρχε αυτή η προτεραιότητα. λοιπόν ε, υπήρχε αυτή η απόφαση στο background. Επίσης τώρα για το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Σωστά είπατε ότι ο πολίτης είναι διοκτήτης των δεδομένων, δηλαδή εγώ ως πολίτης έχω το δικαίωμα να συνδεθώ σε μια θηρίδα, σε μια πύλη και να δω ποιος έχει τα προσωπικά μου δεδομένα και που βρίσκεται το μητρό μου. Έτσι λοιπόν, ε, αν ε, είχα κάποια σχέση με την αστυνομία τις προηγούμενες εβδομάδες, ε, πιθανόν μπορώ να δω αν η αστυνομία έχει αναζητήσει τις προσωπικές μου πληροφορίες στο Μητρό. Αν όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, έχω ούτως ή άλλως το νόμιμο δικαίωμα να κάνω ένα αίτημα, μια ερώτηση στο αρμόδιο θεσμικό όργανο και πρέπει να μου δώσει και μία απάντηση μέσα σε κάποιες ημέρες. Να πρέπει να μου δώσει μία νομικά αιτιολογημένη απάντηση γιατί το όργανο αυτό διερεύνησε τα δεδομένα μου. Δηλαδή, δεν ε, σημαίνει ότι επειδή έχεις πρόσβαση σε κάποια δεδομένα θεωρητικά έχεις και το δικαίωμα να τα δεις τα δεδομένα αυτά. Αυτό είναι ένα ισχυρό μέτρο, δηλαδή αν ε, θεωρείτε ότι αν ε, έχουμε δημόσια τα δεδομένα, ε, μπορούμε να ξαναδώσουμε τον έλεγχο πίσω στον ε, κάτοχο των δεδομένων. Μπορεί στην αρχή δηλαδή αυτή η δημόσια πρόσβαση να φαίνεται ότι δεν είναι ασφαλής, αλλά τελικά αν όλοι γνωρίζουν τα πάντα, καταλήγουμε σε ένα πιο ασφαλές σύστημα. Τουλάχιστον αυτή την οτροπία έχουμε στην Εστονία. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Είναι εμπνευστική, θα έλεγα, όταν βλέπει κανείς ότι έχετε ιδέες και ότι η Εσθονία αντιμετωπίζει πολύ ρεαλιστικά αλλά και με ενθουσιασμό το ζήτημα. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις που θέλω να θέσω. Η Εσθονία είναι αρκετά μικρή χώρα, αν λάβουμε υπόψη τον αριθμό του πληθυσμού και από ό,τι έμαθα το σύστημα βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Είναι πολύ καλό δηλαδή να υπάρχει αυτή η αμοιβή εμπιστοσύνη στην κοινωνία που απλώς αποτελείται από 1,3 εκατομμύρια πολίτες. Εσείς ε, παρουσιάσατε αυτές τις πολύ ρεαλιστικές λύσεις ε, και όταν πήγα στην Εστονία εγώ πάντοτε βλέπω να εμπλέκονται νέοι άνθρωποι αλλά σε ό,τι αφορά τη δομή του πληθυσμού η Εστονία είναι παρόμοια με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λοιπόν η ερώτησή μου είναι πώς ε, μπορεί να ε, αντιμετωπίσετε κάποιους ε, οι οποίοι επιλέγουν πιο αναλογικούς ε, τρόπους, δηλαδή πώς οι άνθρωποι που είναι πιο ηλικιωμένοι, παραδείγματο χάρη, είναι κάπως πιο διστακτικοί να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά σύστημα. Πώς μπορείτε να, να, τους συμπεριλάβετε στο σύστημα. Υπάρχει και κάποιο σύστημα που παράλληλα είναι αναλογικό και ψηφιακό. Εσείς ε, αναφέρατε διάφορους ε, τομείς όπου το σύστημα είναι μόνο ψηφιακό. Αναφερθήκατε το ΣΧΑΡΙ στο Μητρό των Επιχειρήσεων. Ένα άλλο θέμα αφορά την εμπιστοσύνη και τον έλεγχο. Πώς λειτουργεί το όλο σύστημα ως προς το να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσφέρονται πάντα σε αυτούς και στο βαθμό που προβλέπεται και πώς ε, παραδείγματος χάρη συνδέεται, ε, δεν συμβαίνει μάλλον η σύνδεση των δεμένων μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση. Τι κάνετε δηλαδή για να διασφαλίσετε την ασφάλεια, να μην υπάρχει κατάχρηση της εμπιστοσύνης, γιατί παραδείγματος χάρη οι επιχειρήσεις ε, θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα δεδομένα. Θέμα ελέγχου λοιπόν. Τρίτη ερώτηση. Σε σχέση με αυτό το σύστημα της ε, ηλεκτρονικής ε, ε, πολιτογράφησης. Μπορώ να γίνω εγώ, παραδείγματος χάρη, πολίτης ηλεκτρονικά, πολίτης της Εστονίας. Τι ακριβώς προσφέρεται σε αυτό το πλαίσιο. Και σε ό,τι αφορά την εγγραφή των επιχειρήσεων, υπάρχει ο κίνδυνος μια αυστριακή επιχείρηση που δεν της επιτρέπεται πλέον να είναι καταγεγραμμένη στην Αυστρία πολύ εύκολα μέσω του δικού σας συστήματος ε, να πάει στην Εστονία και μετά να επανέλθει στην Αυστρία επειδή θα είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση και θα πληρεί τις προϋποθέσεις στην Εστονία. Δηλαδή, τι κάνετε με το θέμα του ελέγχου του περιεχομένου, αν δηλαδή πληρούνται και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ. Αν με επιτρέπετε να ακούσουμε δύο ακόμη ομιλητέ και έχουμε χρόνο μέχρι τι 10. Μπορείτε να απαντήσετε. Κύριο Φω. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω γερμανικά, αν έχετε την καλή να βάλω τα ακουστικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν και για την παρουσίαση. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ τελικά ήταν αυτό που είπατε ότι ε, ο στόχος μας είναι να ε, δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουν περισσότερα και όχι να περιορίσουμε τα πράγματα. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Αντί να δίνουμε δυνατότητες, περιορίζουμε δυνατότητες. Ε, είναι ενθαρρυντικά αυτά που ακούσαμε λοιπόν. Τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν έχετε ακούσει τις μονοπρόσωπες επιχειρήσεις στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδο μας απασχόλησε αυτό το θέμα και πραγματικά το ζήτημα της ε, κατάχρησης ε, είναι πολύ σημαντικό και για το τομέα της φορολόγησης. Ε, επομένως η ερώτηση είναι κατά πόσον σας έχει απασχολήσει αυτό, έχει παίξει κάποιο ρόλο ιδίως για τις διασυνοριακές επιχειρηματικέ δραστηριότητες. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι κολλήσαμε σε αυτή την προβληματική και δεν είδαμε το πώς μπορούμε να κάνουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε τα πράγματα. Επίσης, την ε, προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το e-privacy, αλλά ε, αυτή η επικοινωνία και αυτά τα μεταδεδομένα για την εφαρμογή των σχεδίων που εσείς αναφέρετε δεν νομίζω ότι μπορεί, είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει εδώ γιατί ουσιαστικά εμείς ε, τα απαγορεύουμε σε ό,τι αφορά τη προσωπικών δεδομένων Πάλι δηλαδή το μυαλό μας δεν κινείται με γνώμα το τι μπορούμε να διευκολύνουμε, τι όδους μπορούμε να ανοίξουμε, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι πώς μπορούμε να προστατεύσουμε, να διαφυλάξουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ περιοριστική αυτή η προσέγγιση. Δεν ξέρω και κατά πόσο λοιπόν συνάδει με το στονικό μοντέλο. Δηλαδή δεν υπήρξαν ε, ε, δεν υπήρχε επεξεργασία σε ό,τι αφορά και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αυτή την προσέγγιση, ιδίω ό,τι αφορά τι μονοπρόσωπε εταιρείε, όπω είπα. Άρα δεν είμαι και τόσο σίγουρο σε ό,τι αφορά την προσέγγιση. Δηλαδή, κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό όπω εσεί το έχετε εδώ παρουσιάσει. Η κυρία Ρέγκνερ επίση είπε πολύ σωστά και προς την ίδια κατεύθυνση ορισμένα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στην πρόσβαση των δεδομένων. Δηλαδή να ξέρετε ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως ε, έκνομα να έχει κάποια πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα. Αυτό δεν μπορούμε να το διευκολύνουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ αν κατάλαβα καλά μπορεί να τα μελετήσει κάποιος, να τα δει και αυτό κάπως καταγράφεται και υπάρχει ένα πρόστιμο, μια κύρωση για όποιον ε, μη εξουσιοδοτημένα ε, είχε πρόσβαση αυτά τα δεδομένα. Τα κατάλαβα καλά όμως ή όχι. Thank you, Mrs. Yeah, thank you very much. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάτι εντυπωσιακό στην Εστονία είναι το εξή. Αν δεν κάνω λάθο, ε, είχατε το προνόμιο να ξεκινήσετε από την αρχή. Ενώ εμείς οι πιο παλιές δημοκρατίες ε, έχουμε δυσλειτουργικά συστήματα και παλεύουμε με αυτά. Έτσι λοιπόν ίσως μπορούμε να αντιλήσουμε κάποια διδάγματα από εσά. Η κυρία Ρέγνερ αναφέρθηκε σε ένα θέμα εμπιστοσύνη Πιστεύω ότι πρέπει να το θυμάμαστε αυτό. Στην Ελβετία υπάρχει πάρα πολύ εμπιστοσύνη προς τους πολίτες ε, και αναπτύσσουν ε, τις ε, πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Έτσι λοιπόν, μήπως αυτό το θέμα του e-residence, της ηλεκτρονικής πολιτογράφησης, θα μπορούσε να οδηγήσει στο να υπάρχει φοροδιαφυγή εταιριών που έρχονται από άλλε χώρε ε, και εγκαθίστανται στην Ιστονία ηλεκτρονικά. Και τι γίνεται με τις ε, κυβερνοαπειλές και το hacking. Ε, φαίνεται ότι είναι τόσο πολύπλοκο όλα αυτά και αλληλοσυνδεδεμένα, επομένως αν συμβεί κάτι πώς το αντιμετωπίζετε. Ναι, αυτές είναι οι ερωτήσεις, επομένως μπορώ να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Έχετε 10 λεπτά να προσπαθήσω να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις για τις πρώτες τέσσερις. Θέμα κοινού και εμπιστοσύνη. Για αυτό που δεν είναι ψηφιακό και πώς το εντάσσουμε. Αυτά που είπα εδώ αφορούν σήμερα και αυτούς που δεν έχουν τρόπο να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές ε, λύσεις αν ας πούμε θέλετε να συστήσετε μια επιχείρηση. Οι πολίτες λοιπόν έχουν πάντοτε δυνατότητα να το κάνουν αυτό με τρόπο παρουσιακό, αναλογικό. Επίσης βλέπουμε καθημερινά ότι όλο και περισσότεροι πολίτες και επιχειρηματίες χρησιμοποιούν αυτές τις λύσεις. Τώρα για την πύλη, για το πόρταλ καταγραφής. Μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων καταγράφονται ηλεκτρονικά στην Εστονία παρά την ύπαρξη δυνατότητα παραδοσιακού τρόπου. Τώρα για τον αναλογικό τρόπο αυτό ανάγεται σε μια δεκαετία πριν όταν είχαμε αυτό το πρόγραμμα που ονομάσαμε το άλμα της τίγρης δηλαδή για αυτούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία Υπήρχαν πολλά προγράμματα σε όλη την Εστονία για να διδάξουν, ας πούμε, στους ηλικιωμένους την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να τους εξοικειώσουν τέλο πάντων με τις τεχνολογικές λύσεις. Τότε αυτό κάναμε. Για το δεύτερο ερώτημα, για τον έλεγχο και την εμπιστοσύνη και την ακαιρεότητα των δεδομένων, αν κατάλαβα καλά. Ρωτήσατε, ας πούμε, πόση πρόσβαση έχουν επιχειρήσει στα δεδομένα. Παρόλο λοιπόν που σας τα παρουσιάσω όλα αυτά ως μία ροή σε ένα-δύο συστήματα τα οποία λειτουργούν στο υπόβαθρο, έχουμε και άλλα συστήματα που λειτουργούν πιο ορατά, όπου εκεί οι τελικοί χρήστες μπορούν να θέσουν δεδομένα τα οποία συνδέονται με αυτά στο υπόβαθρο. Δηλαδή βάζετε τα δεδομένα, ας πούμε τα επιχειρηματικά, αλλά δεν έχετε πρόσβαση στα δεδομένα ε, των ε, βάσεων, δεδομένα, ε, βάσεων δεδομένων για απλούς λόγους όπως η ακαιρεότητα των δεδομένων. Τώρα, αν κάποιος έχει πρόσβαση, ας πούμε οι δικοί μας θεσμοί, στην ίδια τη βάση δεδομένων, τότε έχουμε ένα θέμα διαχωρισμού εξουσιών, απλά και μόνο, και αυτοί που έχουν πρόσβαση στα μεταδεδομένα, σε αυτό το επίπεδο, τότε μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να αλλάξουν κάτι εκεί. Αυτοί όμως δεν έχουν πρόσβαση στα logs, στις καταγραφές, δηλαδή σε όλες τις συναλλαγές, σε όλες τις πράξεις που γίνονται στα δεδομένα. Αυτοί λοιπόν που μπορούν να αλλάξουν δεν έχουν πρόσβαση στα logs, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πάντοτε ένα ίχνος. Αν λοιπόν κάνουμε τα πράγματα ανοιχτά στους επικεφαλείς, ε, βλέπουμε πάντοτε ποιο έχει κάνει τι. Και αυτό διασφαλίζει ότι όσοι έχουν πρόσβαση στα logs, στις καταγραφές, δεν είναι ένα άτομο μόνο, αλλά είναι διάφορα άτομα τα οποία έχουν τις κλίδες τέλο πάντων για πρόσβαση. Αυτό νομίζω μας ευκολύνει και επίσης επιφέρει μια, μια, ένα διαχωρισμό μάλλον των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων για την πρόσβαση. Για, τις, για τους μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους για την πρόσβαση εμείς δεν χρησιμοποιούμε έτοιμες λύσεις Δηλαδή, ναι, τις φτιάχνουμε, τις δημιουργούμε αυτές τις ε, λύσεις και υπάρχουν επιχειρήσει ε, ανάπτυξη λογισμικού που έχουν κερδίσει δημόσιε προμήθειε κτλ. Όμω οι κωδικοί τους επανέρχονται σε εμά στην ε, κυβερνητική πλευρά. του έχουμε εμεί. Αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε αυτοί που συντηρούν το σύστημα, που το λειτουργούν και το διαχειρίζονται. Δεν επιτρέπουν δηλαδή στις ε, Επιχειρήσει τις ε, ιδιωτικέ να αναπτύξουν δικές πρωτοβουλίε όσον αφορά την πρόσβαση και την ασφάλεια. Τώρα για την πολιτογράφηση. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει πολίτης, αλλά πρέπει να συμπληρώσει αυτό το έντυπο, αλλά βέβαια ταυτόχρονα έτσι, στο υπόβαθρο γίνονται διάφορες ε, ενέργειες όπως ένας έλεγχος, ε, διάφορες ενέργειες που αφορούν αυτή την αίτηση. αν ας πούμε πάτε και δείτε την ηλεκτρονική άδεια διαμονής θα δείτε πώς γίνονται όλα αυτά. Τώρα για την καταγραφή, αν μια επιχειρήση ας πούμε στην Αυστρία απαγορεύεται από να, έχει απαγορευτεί από να συναλλάσσεται. Και πάλι είναι το θέμα του τι γίνεται στο όλο αυτό το σύστημα. Έχουμε τους δικαστικούς κλητήρες οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους καταλόγους με υπόψη για τρομοκρατία ή μια μαύρη λίστα τέλος πάντων, ώστε να ξέρουμε ακριβώς ε, τι γίνεται στις διάφορες χώρες της Ένωσης, ώστε να μην μπορούν να μετακινούνται αυτοί οι ύποπτοι ή όσοι βρίσκονται στην ε, μαύρη λίστα. Αυτό το έχουμε ως δυνατότητα στην Εστονία. Μετά, για τη φορολόγηση και τις μονοπρόσωπες εδώ θα έλεγα θα ήταν καλό να δώσουμε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα μας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά πριν το κάνω αυτό να σας πω ότι, όπως είπε η κυρία Χάουταλα, είναι σωστό αυτό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τα κάναμε όλα εμείς από την αρχή. Και αν το κάνετε εσείς αυτό, πάντοτε μπορείτε να τα αλλάξετε. Αντί λοιπόν να αγοράσετε μία έτοιμη λύση που θα μπορούσε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα, δεν μπορείτε να έχετε διασύνδεση με άλλα επικοινωνιακά συστήματα. Έχουμε λοιπόν λύσεις που ενδεχομένω μπορούν να λύνουν ένα πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, να ενταχθούν σε άλλα συστήματα. Εμείς στην Εστονία δεν βρήκαμε κάποιες έτοιμες λύσεις out of the box που θα μπορούσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες μας. Και πιστεύουμε ότι αυτά τα συστήματα τα οποία είναι φτιαγμένα επί τούτου θα μπορούσαν να έχουν διάφορες διαβαθμίσεις και να αντιμετωπίσουν διάφορες αλλαγές ή μεταλλαγές δεδομένων που αλλάζουν γρήγορα. τώρα το λόγο στον κύριο Χάρτμαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που μπορεί να απαντήσει για τα δεδομένα πολύ καλύτερα από εγώ την κυρία Χάρτμαν. Είμαι αναπληρωτή ε, Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Καταρχά, δύο λόγια για την προστασία του δεδομένων. Οι κανόνε είναι οι ίδιοι στην Εστονία όπω στη Γερμανία, γιατί βασιζόμαστε στην κοινοτική νομοθεσία για αυτό το θέμα. Αν λοιπόν μπορούμε στην Εστονία να το κάνουμε νόμιμα, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τα δονομένα νόμιμα, τότε αυτό γίνεται και στη Γερμανία και στην Κροατία και στη Γαλλία, παντού στην Ένωση δηλαδή. Βέβαια, είναι και θέμα εθνικής νομοθεσίας. Αλλά περισσότερο θέμα νοοτροπίας, στην ουσία. Για τη φορολόγηση και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Οποιοδήποτε σύστημα δεδομένων δεν μπορεί πλήρως να αποφύγει τις καταχρήσεις. Βεβαίως, όταν μιλάμε για φορολογική απάτη κλπ, είναι θέμα συνεργασίας μεταξύ φορολογικών υπηρεσιών της Ένωσης και θα έλεγα ότι αν έχετε μία πολύ καλή βάση δεδομένων είναι πολύ πιο εύκολο να ανταλλάξετε δεδομένα με ψηφιακό ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ φορολογικών αρχών γιατί είναι πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό για να καταπολεμήσετε την φορολογική απάτη. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε, κυρία μου, να προσθέσετε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν καλά, αλλά νομίζω τα απάντησα όλα. Για τη ηλεκτρονική διαμονή. Μεγάλο σχέδιο αυτό. Θα μπορούσα να, μιλάω επί 20 λεπτά. Αλλά τέλο πάντων, οποιοδήποτε μπορεί να πολιτογραφηθεί και όταν κάνετε αίτηση, τότε έχουμε αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στο υπόβαθρο, όπως αυτοί που γίνονται όταν κάνετε αίτηση για διαβατήριο. Οι διαδικασίε, αστυνομία, Υπουργείο Εσωτερικών, Δικαιοσύνη τα είναι οι ίδιε όπω με αυτέ τη αίτηση πολιτογράφηση. Αν λοιπόν γίνονται έλεγχοι αφορούν όλα αυτά τα, όλες αυτές τις διαδικασίες και η αίτηση αυτή αφορά μια πενταετία, η οποία μετά θα πρέπει βεβαίω να ανανεώνεται ακριβώς για να δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ελέγχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσω κι εγώ δύο παραδείγματα που μάθαμε στην Εστονία. Γι' αυτά μπορούσε η κυρία Ρέγνερ. για την ηλικία και τη χρήση αυτού του ψηφιακού κόσμου. Μας είπαν, ας πούμε, ότι έχουν και ηλεκτρονικές εκλογές στην Εστονία. Δεν σημαίνει ότι ψηφίζουν ηλεκτρονικά στις εκλογές, αλλά ότι το ηλεκτρονικό σύστημα των εκλογών είναι δίκαιο. Και ένα κύριος που έχει κάνει μια εισήγηση σχετικά εδώ, μας είπε πούμε ότι η φορολογική του δήλωση του έπαιρνε δύο λεπτά στο λεωφορείο μέσω κινητού Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε κατά πόσο ο τρόπος της Εστονίας θα μπορούσε να μεταφερθεί και άλλους άλλες χώρες. Κυρία μου, θέλετε να σχολιάσετε. Ναι, ναι. Για αυτά τα δύο παραδείγματα να πω γιατί υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση σε δύο λεπτά. Επειδή υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διαφόρων μητρών, σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει όλα τα δεδομένα και ως πολίτης απλά και μόνο πρέπει να πατάω ok συνέχεια για να συμφωνήσω με αυτά που βλέπω στην οθόνη. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάμε εκεί γιατί όπως είπαμε στόχος μας είναι η ομαλή λειτουργία. Οπότε αν η κυβέρνηση διαθέτει τα δεδομένα γιατί όχι στο μέλλον να μην ζητάμε μια επιβεβαίωση απλά και μόνο από τους πολίτες. Δηλαδή ο πολίτης ούτε καν θα πρέπει να υποβάλει αίτηση φορολογική γιατί θα, του, θα υπάρχει αυτομάτως συμπληρωμένη από την κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες μου. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Για, ευχαριστώ για τις εισηγήσεις σας. Σας εύχομαι μια ασφαλή πτήση επιστροφής. Εμείς θα συνεχίσουμε με τη δουλειά μας, με τις ψηφοφορίες. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, βγάλτε την καρτούλα σας, και ετοιμαστείτε. Mr. Foss, can we... Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, πόσοι πράσινοι θα ψηφίσουν καταρχάς, γιατί βλέπω τρεις εδώ στην αίθουσα, αλλά μόνο οι δύο μπορούν να ψηφίσουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την έκθεση του κυρίου Μαρίνιου Επίντου. Σχέδιο γνωμοδότησης για την Eurojust. 75 τροπολογία υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 76. Ψήφι υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία Ρίπτεται λοιπόν συμβιβαστική 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Η κάρτα μου. Αλλάξτε. Αλλάξτε μηχάνημα. C'est le même, mais C'est vert, non Ok. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική κάρτα. E Μα πώ δεν ψηφίσαμε με την κάρτα, δεν κάναμε δύο ηλεκτρονικέ επαληθεύσει. Δεν πέρασε η ψήφο μου σε καμία από τι δύο. Ήταν πάντων τουλάχιστον στην πρώτη που ψήφισα κατά και στη δεύτερη που ψήφισα υπέρ. Εντάξει, δεν άλλαξε πάντως ε, η διαφορά των ψήφων ιδιαίτερα. Λοιπόν, είμαστε συμβαστικοί 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Yes. Ναι, έχετε δίκιο. 8. 8 και 82. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Α, καταπίπτει, συγγνώμη. Πού πηγαίνουμε, στην 89. 89 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 10 και 92 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Εγκρίθηκε. Και μία και άλλη. Καταπίπτει 91. Πηγαίνουμε στην 11 και την 93. Ψήφι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 ψήφι υπέρ. Κατά. Θέλω να ελέγξουμε παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 99 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 13 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 100 λέει ο πρόεδρος όχι όχι καταπίπτει συγγνώμη λάθος μου πάμε στην 101 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές απορρίπτεται 14 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 102. Πηγαίνουμε στο τροπολογία 15 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 105. Ψήφι Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Εγκρίθηκε με σαφή διαφορά. Προπολογή 106 ψήφι υπέρ κατά, εποχές, απορρίπτεται. 107 ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 και 108 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 17 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 109 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 111 και 20 ψήφι περ. Κατά. Να ελέγξουμε. has been uh, Εγκρίθηκαν. 114 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 ψήφι περ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 ψήφι περ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ. Απορρίφθηκε. 22 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 116-117 ψήφι υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά αν θέλετε ας το ελέγξουμε να που εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Καλά το είδατε εσείς. Τροπολογή 24. Και... Α, καταπίπτει. Καταπίπτει. Πηγαίνουμε στην 120 ψήφι Εγκρίθηκαν 116 και 117. Yes. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι ψηφίζαμε την τρόπο 24. Δεν την ψηφίζουμε. Αν ψηφίζουμε 116-117, εγώ ψηφίζω κατά. Και αλλάζω το αποτέλεσμα, γιατί ήταν μία ψήφος διαφορά. Θα ήθελα να επαναλάβουμε, παρακαλώ. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία για τις τροπολογίες 116 117. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε βέβαια. And it has been rejected. Απορρίφθηκαν. Με μία ψήφο διαφορά. Που σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 118 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 120 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 25 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ την 25. Εγκρίνεται η 25. 122 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ λέω ότι εγκρίνεται. Αλλά... Α, περνάμε στα 123 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτει 27 27-124 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 125 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126-127 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε. Απορρίφθηκε. «29 και 129. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 128 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130-131 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 30 133 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135 και 137 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 136 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32, 138, 139 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 33 και 140 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 141 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 142 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 ψήφι υπέρ κατά να ελέγξουμε την 144 απορρίφθηκε. 145 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 34 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147, 148 και 149 υπέρ κατά να ελέγξουν παρακαλώ. Απορρίφθηκαν 150-151 ψήφι υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 152 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά ελέγξουμε απορρίφθηκε 156 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 ψήφι υπέρ κατά θα ελέγξουμε Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουν παρακαλώ. εγκρίνεται 162 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 και 163 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 164 ψήφι υπέρ Καταπίπτει δεν καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Ψήφι υπέρ τη 164. Κατά, ποχέ. απορρίπτεται. 40, ψήφι υπέρ. Κατά, Ποχέ. απορρίπτεται. 165, ψήφι υπέρ. Κατά, ποχέ. απορρίπτεται. 166, ψήφι υπέρ. Κατά, Αποχές απορρίπτεται. 41 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167. Α, ήταν ταυτόσιμη, μάλιστα. 168 τότε, ψήφι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. And Απορρίφθηκε 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 170. 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε παρακαλώ. Μάλιστα. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 182 υπέρ ή καταπίπτει πρέπει να καταπέσει είναι η ίδια παράγραφος 181-182 άρα καταπίπτει 43 επομένω Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. Συγγνώμη, 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά εποχές πιθανόν εγκρίνεται αλλά να ελέγξουμε εγκρίνεται στην περίπτωση αυτή 46 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται καταπίπτει 48 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξω Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 καταπίπτει. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε εγκρίνεται Πάμε στην 68 υπέρ κατά Ποχές, Συγκρίνεται. Πάμε στην 67 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Δεν είμαι σίγουρος αν εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Πάμε στην 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 και 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης Άρχεται η ψηφοφορία. We are missing one more. Λείπει ένας ακόμη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαρίνιο Πίντο. Συνεχίζουμε. με την έκθεση Μαστάλκα σε σχέση με την κωδικοποίηση ορισμένων προϊόντων που προέρχονται από την Αμερική, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και το επόμενο, πάλι του κυρίου Μαστάλκα, στατιστικά στοιχεία για τις μεταφορές. Τις και μεταφορές, άρχεται η ψηφοφορία. Ενδιαφέρεται κάποιος άλλος να ψηφίσει. Μας λείπουν τρία άτομα που δεν έχουν ψηφίσει. Ωραία. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Μαστάλκα. Και εδώ ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες.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 Κυρία Χαουτάλα, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να είχαν μείνει λίγο περισσότεροι συνάδελφοι, γιατί είναι κάπως ε, έκτακτη κατάσταση με τις επιγραμμικές ε, πωλήσει ε, υλικών αγαθών και επειδή ο κύριος Φως είναι εισηγητής ενός αδελφικού χαρτοφυλακίου που αφορά τις επιγραμμικές πωλήσει ε, προϊόντων με ψηφιακό περιεχόμενο. Εδώ και ένα χρόνο εργαζόμαστε επί δύο προτάσεων που συνδέεται με την ψηφιακή ενιαία αγορά, επιγραμμική αγορά ψηφιακών προϊόντων, επιγραμμική πώληση συγγνώμη, και επιγραμμική πώληση ε, υλικών ε, προϊόντων, παραδείγματος χάρη πλυντήρια. Όταν αρχίσαμε με αυτά τα υλικά αγαθά και εγώ είμαι η συγγήτρια σε αυτή την επιτροπή Βάση του άρθρου 54, ενώ το άρθρο 55 καλύπτει το ψηφιακό περιεχόμενο, Νίκο και Τζούρι λοιπόν, εκεί είναι σε ίση βάση. Όταν ε, ξεκινήσαμε ε, όλη τη διαδικασία με την ανακοίνωση refit της Κομισιόν, ξεκαθάρισαν ότι βάσει του Refit ε, είχαν προτείνει να ε, διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής ε, της πρότασης και σε πωλήσει offline, πέρα από τις επιγραμμικές πωλήσει των υλικών αγαθών. Όμως είναι σημαντική αυτή η αλλαγή, θα έλεγα. Όταν προσπάθησα να πω ότι βάσει της καλύτερης νομοθεσίας η Κομισιόν θα έπρεπε να κάνει τη μελέτη αντικτύπου της επέκτασης του πεδίου εφαρμογή ε, από τις online στις offline πωλήσει. Νομίζω ότι υπήρχε ευρεία συμφωνία. Εγώ δεν ε, συμφωνούσα ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει αυτή τη μελέτη αντικτύπου, ενώ κανονικά η Κομισιόν θα έπρεπε να κάνει τη μελέτη αντικτύπου και να έρθει με μία τροποποιημένη πρόταση. Εμείς ε, λοιπόν εργαστήκαμε επί του θέματος αυτού και επί των δύο προτάσεων, τις επιγραμμικές πωλήσει ψηφιακών προϊόντων και τις επιγραμμικές πωλήσει υλικών αγαθών. Συνεργαστήκαμε στενά και το ίδιο ισχύει και για τις δύο επιτροπές. Τώρα όμως ξέρουμε και μόνο άτυπα το γνωρίζουμε αυτό, ίσως βέβαια η γραμματεία να έχει λάβει μια επίσημη ενημέρωση από την Κομισιόν ότι μετά από ένα έτος ε, επιστρέφουμε και πάλι στο μηδέν. Δηλαδή η Κομισιόν πιθανότατα κατόπιν συμβουλής του Συμβουλίου αποφάσισε να παρουσιάσει μια τροποποιημένη πρόταση με διεύρυνση του πεδίου και στις ε, offline πωλήσει Και τι να πω τώρα, τα έλεγα. Έπρεπε να έχουμε ζητήσει στην Κομισιόν ε, να κάνει τη δουλειά της τότε όπως έπρεπε και τώρα εξακολουθούμε να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν για το τι ακριβώς θα κάνουν. Όμως, από έχω καταλάβει, στα τέλη του μήνα η Κομισιόν θα αποφασίσει για μια τροποποιημένη πρόταση και ελπίζω να έχει και μια μελέτη αντικτύπου και να μην μείνουμε σε αυτή που κάναμε εμείς ε, για αυτούς, εξ ονόματός τους. Τώρα, δεν υπάρχουν ε, και πάρα πολλά άρθρα που να ε, διέπουν το τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Η Κομισιόν μπορεί να ξαναστείλει την πρότασή της και πάλι στο Κοινοβούλιο. Κοιτάζω εδώ το άρθρο 63 και ίσως το εδάφιο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στην κατάσταση να είναι ότι η Κομισιόν μπορεί να ξαναστείλει την πρότασή της στο Κοινοβουλίο κατόπιν αιτήματος της Αρμόδιας Επιτροπής όταν η φύση του προβλήματος, ε, όταν μιλάμε για ουσιαστικές αλλαγές, ή αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Όμως κανένα εδάφιο δεν λέει ε, ότι στην περίπτωση που η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της και σκοπεύει τώρα να την κάνει. Τέλος πάντων, εδώ βρισκόμαστε και φυσικά δεν πρέπει να πάμε πάλι στο μηδέν, γιατί είχαμε διευρυμένες συζητήσεις για ιδιαίτερα πολύπλοκες πτυχές της αρχικής πρότασης, έχοντας κατά νου ότι το πεδίο εφαρμογή θα μπορούσε πράγματι να διευρυνθεί. Γιατί δεν έχει νόημα να έχουμε διαφορετικούς κανόνες για επιγραμμικές και μη επιγραμμικές πωλήσει. Αυτό είναι σαφές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το έργο ε, για την ε, πρόταση επί της οποίας είναι αρμόδιος ε, ο κύριος Φως για τα ψηφιακά, δηλαδή το ψηφικό περιεχόμενο, έχει προχωρήσει πιο πολύ. Νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και στο Συμβούλιο και πιστεύω ότι και οι σκιώδεις εισηγητές μαζί με τον κύριο Φως και τον κύριο Γκέπχαρτ από την πλευρά της Επιτροπής ΙΜΚΟ έχουν φτάσει κοντά σε τελικές λύσεις δεν είναι ακόμα εκεί, αλλά από ό,τι κατάλαβα η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στη μεικτή συνεδρίαση των Επιτροπών αυτό το μήνα. Σωστά, σωστά κύριε Φως. Ωραία. Όμως ε, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο με την πρόταση για τελικά αγαθά. Καταρχήν, ε, είναι σωστό να περιμένουμε την τροποποιημένη πρόταση και να δούμε τι ακριβώς θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν, η πρότασή μου είναι επειδή μας λείπει κάποια καθοδήγηση, να συζητήσουμε αν θα θέσουμε νέα προθεσμία για υποβολή τροπολογιών και αν θα έχουμε νέες ε, διαπραγματεύσεις για συμβασμό και αν θα επανέλθει η πρόταση στην Επιτροπή το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Και όσοι θέλουν να ευθυγραμμίσουν αυτές ε, τις δύο οδηγίες, ίσως να μην ήταν αυτό η ιδανική λύση. Αλλά τώρα έχουμε κατανοήσει καλά ποια στοιχεία μπορούν να ευθυγραμμιστούν και ποια δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν. Λόγω έλλειψης κοινών χαρακτηριστικών, επειδή μιλάμε για διαφορετικά είδη προϊόντων. Εγώ προτείνω λοιπόν να περιμένουμε την τροποποιημένη πρόταση και ελπίζω ότι και η Επίτροπος Γιούροβα θα έρθει να την παρουσιάσει εδώ ίδια και κατόπιν να θέσουμε νέα προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και για να έχουμε νέες διαπραγματεύσεις. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα με αυτό, γιατί και το Συμβούλιο τώρα αρχίζει τη συζήτησή του επί της πρότασης αυτής για τελικά υλικά αγαθά. Το κύριο θέμα που πρέπει να λύσουμε είναι το επίπεδο της εναρμόνισης. Έχουμε ουσιαστικά ένα δύσκολο ιστορικό στο ευρωπαϊκό δίκαιο καταναλωτών γιατί ουσιαστικά ε, έχει να κάνει με ουσιαστικά στοιχεία του δικαίου αυτού και πολλοί αισθάνονται ότι το κοινοβούλιο δεν θα είναι αυτό που θα περιορίσει και θα μειώσει τα δικαιώματα των καταναλωτών σε κάποιες χώρες. Υπάρχουν αποκλήσεις, όμως θα πρέπει να στοχεύσουμε σε ψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κάποια ελάχιστη εναρμόνιση με πολύ καλά προσδιορισμένες ε, πτυχές, πού στοχεύουμε δηλαδή και σε ποια σημεία εναρμονίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να λύσουμε όλο αυτό το ζήτημα. Okay. Uh, well, thank Ευχαριστώ για τη δήλωσή σας. Ο κύριος Φως έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα, αλλά παρακαλώ αν θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Χάιντι Χάουταλα εξέθεσε ουσιαστικά το πρόβλημα και μάλιστα με πολύ εύγλωτο τρόπο. Ουσιαστικά και στις δύο επιτροπές, την Επιτροπή Γιούρι και την Επιτροπή Ίμκο, έχουμε το εξής ζήτημα. Είναι μεν πολύπλοκο, αλλά το θέμα σε όλες τις περιπτώσεις και αυτές που αναφέρεται υλικά αγαθά, ψηφιακά, αγαθά αλλά εντάσσονται ουσιαστικά σε μια βασική ιδέα. πρέπει να κινηθούμε παράλληλα και στις ε, περιπτώσεις, σε τέσσερις περιπτώσεις ε, και σε ό,τι αφορά την ε, μελέτη αντικτύπου αυτό που είπα. Τώρα έρχεται αυτό το επόμενο βήμα. Έχουμε άλλη μια διακοπή με αυτή την τροποποιημένη πρόταση και μας δημιουργεί ανασφάλεια για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, δηλαδή στον τομέα το ψηφιακό εμείς προχωράμε και προσπαθούμε και με τις... Ε, ε, με τις συναδέλφους που ασχολούνται με την οδηγία για τα υλικά αγαθά να συντονιστούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι κανόνες ε, οι οποίοι θα συμφωνήσουμε δεν θα πρέπει μετά να μην έχουν κανένα νόημα. Δηλαδή από διαδικαστικής άποψης θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για να μην διαφοροποιηθούμε σε σχέση με το τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. διότι πιστεύω ότι και από πλευράς περιεχομένου και από πλευράς λογικής καλό είναι να υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ δηλαδή των ε, υλικών και μη, ε, και μάλλον συγγνώμη των επιγραμμικών και μη επιγραμμικών πωλήσεων. Θα πρέπει από την αρχή να γίνει αυτό. Πράγματι υπάρχει το ζήτημα της εναρμόνισης ε, και για τους δύο τομείς ε, που δεν αντιμετωπίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά αν μπουν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία ε, δικαιολογούν ε, την καλύτερη εναρμόνιση, θα πρέπει να δούμε μετά κατά πόσον θα υπάρχουν ε, διαφορές ή όχι. Αλλά νομίζω ότι προς το παρόν είμαστε σε καλό δρόμο. Ερώτηση προς την κυρία Χάουταλα. Λέμε να ψεφίσουμε στην ΙΜΚΟ μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, έτσι. Δεν είμαι βέβαιη, λέει η κυρία Χάταλα. Το συζητάνε οι γραμματείες. Βλέπω όμω ότι ο κύριος Άρημα, το εισηγητής στην ΙΜΚΟ, φαίνεται να θέλετε να προσαρμοστεί στην κατάσταση. Βλέπει ότι τροποποιούμε την πρόταση. Θα ήταν ρεαλιστικό αυτό νομίζω, σε περίπτωση που υιοθετήσει η Κομισιόν την τροπομένη πρόταση μέχρι το τέλος του μήνα. Αλλά κάπως είμαστε στο άγνωστο, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα επίσημα σχεδιάζει να κάνει η Κομισιόν. Πρόεδρος. Αλλά περιμένουμε την ΙΜΚΟ, έτσι. Ναι, και εμάς περιμένουμε. Νομίζω υπάρχει φιλική συνεργασία. Γιατί ο κανόνας 54 δίνει στην Επιτροπή μας ισχυρή θέση, όχι 55, αλλά και ο 54 μας δίνει μια ισχυρή θέση. Πρόεδρος. Να γράψω στον πρόεδρο του για να διευκρινίσουμε τα πράγματα, κύριε Χάτελα. Ναι, νομίζω σήμερα θα το ρυθμίσουν ούτως ή άλλως οι γραμματείες. Αλλά ναι, σε δεύτερη φάση βέβαια. Ο κύριος Φως. Ίσως για να προσπαθήσω να τα διευκρινίσω κάπως τα πράγματα. Έχουμε την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και έχουμε θέσει ψηφοφορία την αναβολή. Δεν ξέρω. Για τέλη Νοεμβρίου. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορούσε να συνδυαστεί και με τα υλικά αγαθά. Εμείς το συζητήσαμε, δηλαδή πόσο θα μας κοστίσει αυτή η χρονική αναβολή, να το αναβάλουμε για την Πέμπτη και επειδή υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, εξωτερικές δράσεις, εμείς είπαμε ότι θα το αναβάλουμε για τέλη Νοεμβρίου, σε ό,τι αυτό το ψυχιακό περιεχόμενο. Αλλά για τα υλικά αγαθά δεν ξέρω ακριβώς ε, τι μπορείτε να κάνετε, θα μπορείτε να το έχετε ολοκληρώσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ναι, κυρία Χαουταλά. Ναι, παρακαλώ. Άλλη μια διευκρίνηση. Από ό,τι κατάλαβα και μπορεί να το επιβεβαιώσει, να το διευκρινίσει ο κ. Φως, η στενοκή Προεδρία με ενθουσιασμό ήθελε να ολοκληρώσει τον τριμερή διάλογο κατά διάρκεια της Προεδρίας τους για αυτή την πρόταση. Ίσως λοιπόν είναι ακόμα δυνατό, πάνε κάπω θαύμα βέβαια, αλλά τέλο πάντων αυτό θέλουν να πετύχουν, ένα θαύμα. Και η Κομισιόν δεν ευχαριστήθηκε και τόσο ότι όταν έμαθε ότι δουλεύαν πάνω σε αυτή την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο. Πάντως μπορούμε να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε δύο προτάσεις. Πάντως δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αν δεν συμφωνήσουμε για το ποια στοιχεία θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και ποια δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν, και έχουμε διαφορές γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το Συμβούλιο μόλις ξεκίνησε τη δουλειά για τελικά αγαθά, μπορούμε να χρειαστούμε να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω χρόνο. Πρόεδρος, ναι, θα στείλω μια επιστολή στον πρόεδρο της ΣΥΜΚΟ για να ζητήσουμε κάποιες διευκρινήσεις μετά από αυτά που συζητήσαμε εδώ. Ελπίζω αυτό να αρκεί προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με το θέμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, σημείο 21. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραβίασης των Δικαιωμάτων Διανοτικής Ιδιοκτησίας ο λόγος του κύριο Καβαντά που είναι και μέλος εκεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ταχύτατα για να πάμε γρήγορα. Όπως ξέρετε, 26-27 Σεπτέμβρη έγινε η ετήσια ολομέλεια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησία. Είχαμε γύρω στου 100 συμμετέχοντε από όλε τι χώρε μέλη βέβαια, από τον ιδιωτικό τομέα, τον ενδιαφερόμενο, κοινωνία πολιτών και άλλους. Να τονίσω ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να σας μεταφέρω, το άρθρο 8 του 386 του 12 δηλαδή η παρουσίαση πρώτων στοιχείων αξιολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την Γενική Διεύθυνση Grow της Κομισιόν. Αυτό το άρθρο του κανονισμού έχει ως στόχο να εξεταστεί λεπτομερώς ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και να απευθυνθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις. Πρέπει κάποια πράγματα λοιπόν εδώ να γίνουν. Τα προκατακτικά αποτελέσματα που μας παρουσιάστηκαν ήταν πολύ θετικά και ο ρόλος του παρατηρητηρίου εκτιμάται ιδιαίτερα. Να το τονίσω αυτό. Και ήμουν ο μόνος ευρωβουλευτής που πήγε αυτήν την ολομέλεια. Καταλήγοντας, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο θα πρέπει να έχει ενισχυμένο ρόλο σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Θα ήταν καλό επίσης το παρατηρητήριο να είναι σε θέση να ενισχύσει οικονομικά τις διάφορες δράσεις σε εθνικό επίπεδο με τη συνεργασία της Europol και τρίτον να κάνω μια παρατήρηση το παρατηρητήριο δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε μια αρχή εφαρμογής αλλά θα πρέπει να αντίθετα να αναπτύξει τις δυνατότητες συντονισμού των εθνικών αρχών που έχουν αυτή την αρμοδιότητα όσον αφορά την καταπολέμηση των παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοική ιδιοκτησία. Ένα φαινόμενο που γίνεται όλο και πιο έντονο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Σχόλια από τα μέλη. Δεν βλέπω κάποιον. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημείο 22. αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Εγώ είμαι ο συγητής Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για τις τροπολογίες που καταθέσατε στο φάκελο αυτό. 59 έλαβα τροπολογίες που διάβασα προσεκτικά και που θα λάβω υπόψη μου δεόντως για τη σύνταξη τελική γνωμοδότηση Να αναφερθώ σε κάποιες από τις πιο σημαντικές τροπολογίες και τα θέματα που έφυγαν Συγκεκριμένα, η επαναδιοχέτευση που αφορά τις περιπτώσεις δέσμευσης και δίμευσης. Πολλοί συναδελφοί τονίζουν την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών και τρίτων χωρών και μεταξύ των διαφορών αρμοδίων αρχών στις χώρες μέλη. Μιλούν επίσης για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας, ουσιώδες ζήτημα όσον αφορά την θέσπιση ενός ενιαίου προτύπου που αφορά τις δεσμεύσεις και τις δημεύσεις. Επίσης, απαιτείται η άμεση αναγνώριση αυτών των ενταλμάτων δέσμευσης και δήμευσης και επίσης είναι απαραίτητη μια διαδικασία ομοιόμορφη όσον αφορά την εκτέλεση αυτών των ενταλμάτων. Πάντοτε βέβαια σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης. Άλλο ένα ζήτημα για το οποίο κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες και το οποίο σχετίζεται με τις δυνατότητες προσφυγής όσον αφορά τις αποφάσεις δέσμευσης και δίμευσης συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στον φάκελο και στις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους οι αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις προτάσεις σας λοιπόν, ο Πρόεδρος, να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 21 του Νοέμβρη. Αυτά από μένα, η κυρία Κάφμαν νομίζω θέλει το λόγο. Ναι, πράγματι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και για τον τρόπο με τον οποίο συνοψίσατε και παρουσιάσατε τις τροπολογίες, αλλά και βέβαια για το έργο που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση αυτή θα είναι μια πολύ καλή γνωμοδότηση η οποία θα προκύψει από τη συνεργασία μας. Ε, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, διότι τα περιουσιακά στοιχεία, τα χρήματα, τα οποία ε, δημιουργούνται με παράνομες δραστηριότητες, ε, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να παραμείνει στα χέρια των εγκληματιών και να μπορούν με αυτό τα χρήματα να προχωρήσουν σε νέες τέτοιες παράνομες δραστηριότητες, διότι από ό,τι φαίνεται το πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων αυτών, ε, το 98% δεν ε, το κατάσχουμε και γι' αυτό είναι πολύ καλό αυτό το εργαλείο το οποίο έχει προτείνει η Κομισιόν, δηλαδή έναν κανονισμό για την απλούστευση του νομικού πλαισίου που ισχύει μέχρι τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη διάταξη ό,τι αφορά την πληροφόρηση, να είναι πιο μικρές αλλά σε οι προθεσμίες, ε, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρχών στον τομέα αυτό. Επίσης ότι οι θυγόμενοι θα πρέπει να μπορούν να ε, λαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και εποπτείας ό,τι αφορά τις ε, διάφορες ε, νομικές πράξεις και τις εντολές. Τι γίνεται όμως με αυτά τα αγαθά, τα περιουσιακά στοιχεία ε, τα οποία δημεύονται ή δεσμεύονται. Αν υπάρχει δηλαδή από το ένα κράτος μέλος μια άλλη, μάλλον δέσμευση περισσότερων στοιχείων που σχετίζονται με ένα άλλο, τι γίνεται με αυτά και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το που δημιούργησαν ε, ζημία αυτές οι παράνομες δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε με τη συνεργασία μας, όπως είπα, να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες παρατηρήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω εγώ, Πρόεδρε, για τη δουλειά που κάνατε κατέθεσα τρει τροπολογίες και ελπίζω να τι περιλάβετε στην πρότασή σας. Όσον αφορά δηλαδή τι δημεύσει προ και θα πρέπει να τι εξετάσουμε προσεκτικά. Επίσης μιλάω και για την διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ αρμοδίων αρχών. Οπότε προσβλέπω στην τελική πρόταση εκ μέρου σα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Μήπω η Κομισιόν επιθυμεί το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Οπότε. Τελειώσαμε και με το 22 και νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει την πρωινή ημερήσια. Όχι, λέει ο λάθος, λάθος. Ε, Έχουμε και άλλα να κάνουμε. 23, σημείο 23. Ετήσιες εκθέσεις 15-16 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Η κυρία Ντελβό, η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πολύ σύντομα γιατί ήδη κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή. Φέτος δεν είναι ετήσιες εκθέσεις, αλλά διετής. Γιατί το 15 και το 16 πάνε μαζί. Και όπως πάντα θα πρέπει να αναζητήσουμε μια ισορροπία μεταξύ... Πώς να το πω, πώς να το πω. να αναζητήσουμε το πιο αποτελεσματικό επίπεδο ώστε να προωθήσουμε τις πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις αρχές της επικορικότητας και της αναλογικότητας που είναι πολύ σημαντικές για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και θα έπρεπε να μας διευκολύνουν ώστε οι πολίτες, τα εθνικά κοινοβούλια, τα περιφερειακά κοινοβούλια να συμμετέχουν και να δείξουν ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και όχι να αποτελούν ένα φραγμό για την ε, εξέλιξη των ευρωπαϊκών κειμένων. Για τις εκθέσεις λοιπόν αυτές, ιδιαίτερα για την έκθεση του 2015, η Κομισιόν θέτει το πακέτο Better Regulation με γραμμές κατευθυντήριες για την αξιοποίηση της υπερκουρικότητα και της αναλογικότητας και διαβάζοντας την αξιολόγηση αντικτύπου που έγινε IB και μετά έγινε SRB διαπιστώνω ότι η Κομισιόν πράγματι καταβάλει προσπάθειες λέγοντας ας πούμε για το 2015 ότι 23% της αξιολόγησης αντικτύπου χρειάζεται βελτίωση και το 16 μόνο 16%. Οπότε βλέπετε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά πάντοτε μπορούμε να βελτιωθούμε. Να υπενθυμίσω επίσης ότι και η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι επιθυμητή σε διάφορα επίπεδα πρόσβαση μέσω ΣΔΡΕΦΙΤ στις αξιολογίες αντικτύπου, συμμετοχή στις διαβουλεύσεις. Υπάρχει στο σελίδα της Κομισιόν που ξεκίνησε το 2015 και που περιορίζει τα διαδικαστικά για την έκφραση των πολιτών και των βουλευτών και επίσης η περιφέρεια των συγγνώμη, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει μια ομάδα 12 πυρογνωμών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας. Αναφέρω λοιπόν αυτά τα υπάρχοντα εργαλεία στην έκθεσή μου. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και πιο προσεκτικοί και επικοδομητικοί γιατί ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μια ομάδα, τη συγκρότηση μιας ομάδας η οποία ακριβώς θα ασχοληθεί με την επικορικότητα και την αναλογικότητα. Και με ανυπομονησία αναμένουμε την συγκρότηση αυτής της Task Force για αυτά τα δύο ζήτηματα. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές που θα εφαρμόσω κατά τη σύνταξη της έκθεσης για το χρονοδιάγραμμα. Το Νοέμβριο θα το υποβάλω και μετά το Δεκέμβριο επίσης και μετά ελπίζω να ψηφίσουμε τον να Βάρη στη ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Σκιώδης από το ΕΛΚ ε, θα ήθελε να εκφράσει την άποψή του για την γνωμοδότηση αυτή ε, και τα, θα τα διαβάσω εγώ. Η κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριοι συνάδελφοί, μα αναγκάζει να θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εύρωστη νομοθεσία ώστε να μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και να υπάρξει προστέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο που έφερε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ήπειρό μα. Οι πολίτε μα δεν θέλουν μια Ευρώπη που θα χάνεται στι λεπτομέρειε. Μια Ευρώπη θέλουν που θα αγωνίζεται εκεί που μπορεί να γίνει διαφορά και γι' αυτό χρειάζεται μία διευκρινήση των διαχωριστικών δραμμών μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη ε, και από τις εθνικές αρμοδιότητες για καλύτερη εφαρμογή των αρχών της επικορικότητας και της αναλογικότητας. Έτσι λοιπόν να χαιρετίζω την έγκριση από το Μά, το του του πακέτου καλύτερη νομοθεσία από την Επιτροπή και του νέου μηχανισμού διαβούλευσης και ανατροφοδότησης, feedback. Lighten the Load ε, είναι ε, ε, μια πρωτοβουλία της Κομισιόν στο και έχουμε και την πλατφόρμα Refit από το 2016. Και τα δύο αυτά εργαλεία δίνουν στους εμπλεκόμενους φορείς δυνατότητα να έχουν επικοινωνία με την Κομισιόν για, κατα... για... για ρυθμιστικά μέτρα τα οποία θεωρούν υπερβολικά έχουμε την διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία που εγγράφει τον Απρίλιο το 2016. και αυτή δείχνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα είναι προσιλωμένα στο στόχο της καλύτερης νομοθεσίας. Ε, τα εθνικά κοινοβούλια στο ρόλο τους ως εκπρόσωποι των πολιτών σε εθνικό επίπεδο έχουν να διαδραματίσουν και αυτά σημαντικό ρόλο για την ε, υπέρβαση των διαφορών μεταξύ κοινή γνώμη και ε, δημόσιο τομέα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ των αριθμών των αιτιολογημένων γνωμών που επιβλήθησαν το 2015 και το 2016. Από 864, σημαντική αύξηση που δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια αρχίζουν να δραματίσουν έναν όλο και πιο ενεργό ρόλο στην έγκριση ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τέλος, θέλω να δώσω έμφαση στο εξής. Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της χάρξης πολιτικής για να φανεί κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πετύχει καλύτερα τους στόχους από το τοπικό ή το περιφερειακό ε, ή το εθνικό επίπεδο. Ελπίζω με τις δύο προτάσεις να έχουμε καλύτερη νομοθεσία. Άρα δεν υπάρχουν βέβαια προβλήματα. Οι πολίτες έτσι θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ με την κυρία Ντελβό και ελπίζω να συνεχιστεί η εξαιρετική συνεργασία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, ευχαριστώ κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Τελβό που ανέλαβε αυτό το έργο για την επικουρικότητα και την αλογικότητα για τα 15 και 16. Είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των δύο ετών. Εγώ, όπως ξέρετε, ε, ακολουθώ ιδιαίτερα την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά τις αρμοδιότητες στην Ένωση. Έχω όμως κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την τήρηση, του σεβασμό της επικουρικότητας. Τα έγγραφα που υπάρχουν επιβεβαιώνουν αυτή την απόψη μου, γιατί έχουμε μόνο τα στοιχεία ο αριθμό των ανακοινώσεων, α πούμε, των Εθνικών Κοινοβουλίων το 2015 και το 2016. Βλέπουμε ότι έχουμε 254 ανακοινώσει των Εθνικών Κοινοβουλίων το 2015 και 410 το 2016. Και αν δούμε τις λεπτομέρειες θα δούμε ότι το 2015 είχαμε 8 ανακοινώσει, οι οποίες ήταν γνώμε τεκμηριωμένες και το 2016 ήταν 116. Είχαμε μια τεράστια λοιπόν αύξηση και όπως ο κύριος Βος μπορεί κανεί να είναι αισιόδοξο, γιατί μπορεί να σημαίνει ότι τα εθνικά κοινοβούλια τέλο πάντων συμμετέχουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, αλλά δεν έχω εγώ την ίδια ερμηνεία. Κάθε άλλο, τα εθνικά κοινοβούλια βλέπω ότι ενοχλούνται από την παρέμβαση της Ένωσης στους τομείς αρμοδιότητά τους και γι' αυτό κάνουν τις ανακοινώσεις. Εγώ θεωρώ δυστυχώς ότι η επικουρικότητα τηρείται όλο και λιγότερο και παρά τις υποσχέσει για καλύτερη νομοθεσία, νομίζω ότι αντί λοιπόν να φύγουμε προς τα μπρος, βλέπουμε ότι έχουμε παράκαμψη της επικουρικότητα και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αδίαιο έξοδο. Ελπίζω να κάνω λάθο. Ελπίζω η κυρία Ντελβό να μου αποδείξει ότι κακώς ερμηνεύω αυτά τα στοιχεία, αλλά νομίζω δυστυχώς έχω σοβαρές εμφωλίες. Κυρία Αντελφού, κύριε Λεμπρετών, τι έργο μου θα είναι δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι οι παρεμβάσεις αποδεικνύουν ακριβώς τη διπλή φύση των ε, θεμάτων της επικριτικότητας και της αναλογικότητας. Δηλαδή, μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με θετικό μάτι και να πούμε ότι είναι πολύ καλό που εμπλέκονται τα κοινοβούλια και κάνουν μεμοδοτήσεις. Εγώ αυτή την ερμηνεία κάνω, τουλάχιστον για τα κοινοβούλια τεχνικά που ξέρω, που γνωρίζω καλά, ή μπορούν να πούν, να πει κανεί ότι αρνητικά, απεσιόδοξα και να πει κανεί ότι αυτό είναι κακό σημάδι. Πάντως μου βάζετε μια πρόκληση κύριε Λεμπρετών. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι ότι είμαι ε, στο, σίγουρη ότι είμαι στο ύψος του περιστάσεων, αλλά πάνω θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποκριθώ. Ναι. Και εγώ μάλλον συμμερίζομαι την θετική προσέγγιση γιατί νομίζω ότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η σύνδεση μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και ο αυξανόμενος αριθμό εδώ αποδεικνύει ακριβώ το ότι τα εθνικά κοινοβούλια αρχίζουν να ενδιαφέρονται για αυτά που κάνουμε εμεί εδώ. Οπότε εγώ το ερμηνεύω θετικά. Θεωρώ ότι είναι θετικό αυτό το στοιχείο. Ωραία. Ο κύριος Καβαντά. Ναι. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και η τροπή της. Κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνείτε ή αν συμφωνεί και ο κύριος Λεμπερτών, θα του απονείμω το τριμηνιαίο μετάλλιο του απεσιοδόξου τιμής. Ναι, πολύ καλή πρόταση λέει ο πρόεδρο. μπράβο. Μήπως η Κομισιόν επιθυμεί το λόγο για αυτό το θέμα. Παρακαλώ Κομισιόν. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση σε σχέση με τις στατιστικές που ανέφερε ο κύριος Λεμπερτών και εμείς τις έχουμε και παρατηρούμε μια τάση ότι πριν και μετά την αλλαγή της εντολής έχουμε κάποια αλλαγή σοβαρή σε σχέση με τον αριθμό των γνωμοδοτήσεων από τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί ακριβώς έχουμε νέε προτάσεις από την Κομισιόν. Οπότε το να ερμηνεύει κανείς στοιχεία απόλυτα σε σχέση με τις γνωμοδοτήσεις, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται προσεκτικά. Και μία παρατήρηση για την Task Force που προανήγγειλε ο κύριος Γιούνκερ στην ομιλία του. Αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν εργαζόμαστε πάνω στις μεθόδους εργασίας και στις λεπτομέρειες για αυτή την Task Force. Όπως είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, θα αποτελέσει μια ευκαιρία για τα Εθνικά και, και το Ευρωκοινοβούλιο να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία όπου η Κομισιόν θα προσπαθήσει να εντοπίσει σε μεγαλύτερο μικρότερο πλαίσιο τα σημεία όπου οι δραστηριότητες μπορεί καλύτερα να βρίσκονται σε τοπικό αντί για ευρωπαϊκό επίπεδο ή αντίστροφα. Εμείς λοιπόν συμμετέχουμε ενεργά στην συγκρόση αυτή τη Task Force με στόχο να υλοποιηθεί πλήρω και να είναι ενεργή φέτο. Και βεβαίω όταν ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες μας θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για αυτές τις πληροφορίες. Χαίρομαι να δω ένα αποτέλεσμα του έργου αυτής της εργασίας της Επιτροπής, γιατί όλοι συμφωνούν ότι κάποιες αρμοδιότητες θα μπορούσαν να επιστραφούν στα κράτη-μέλη, αλλά όταν ε, γίνεται η συζήτηση σε σχέση με το ποιες αρμοδιότητες δεν υπάρχουν απαντήσεις. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Συνεχίζουμε με το σημείο 24. Έλεγχος ε, κατά κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και λοιπόν εκτελεστικών μέτρων. Ο κύριος Λεμπρετών είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα που ήδη σας έχω παρουσιάσει. Πρόκειται με τη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν εξελιχθεί. Είναι αρκετά τεχνικό το ζήτημα. Είμαστε αρμόδιοι σε σχέση με το άρθρο 66 του ιστορικού κανονισμού του Κοινοβουλίου για να δούμε τις εκτελεστικές πράξεις, να τις ελέγξουμε. Εγώ δεν είδα να υπερβαίνει κάτι τις αρμοδιότητες της Κομισιόν μέχρι τις 4 Οκτωβρίου ήταν η προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων. Καμία αντίρρηση δεν υποβλήθηκε. Έτσι λοιπόν μπορώ να σας πω ότι η άποψή μου φαίνεται να εγκρίνεται από όλου. Τίποτα δεν υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Όλα πάνε καλά λοιπόν. Για μια φορά να δεν είμαι και πάντοτε απεσιόδοξος. Μάλιστα, με εκπλήσετε, κύριε Λεμπρετών. Πολύ ωραία. Παρατηρήσει για το 24. Αν όχι, να περάσουμε στο 25. Ο κύριος Καβαντά είναι ο εισηγητής. Λοιπόν, 25 και 26, τα σημεία αυτά θα τα σχολιάσω εντάχει. Πρόκειται για το θέμα των εκτελεστικών πράξεων ε, σε ό,τι αφορά θέματα περιουσιακών ε, σχέσεων ε, των ζευγαριών με καταχωρημένη συμβίωση και των συζύγων σας εστάλει ένα έγγραφο από τη γραμματεία για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από τους συναδέλφους βουλευτές ε, ως την προθεσμία που είχε τεθεί από τη γραμματεία της Επίτροπής μας. Έτσι λοιπόν τα προσχέδια των εκτελεστικών πράξεων συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης ε, και δεν υπερβαίνουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, δεν θα έπρεπε να θέσει καμία αντίρρηση για την υιοθέτηση αυτών ε, των προσχεδίων. Και εδώ ολοκλήρωσα το σημείο αυτό. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα σημεία 25 και 26 από κοινού. Υπάρχουν παρατηρήσεις από τους συναδέλφους. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος το λόγο. Λοιπόν, σημείο 27, άρθρο 42 για την επικουρικότητα. Εδώ απλώς ε, σημειώνουμε ότι έχουμε λάβει δύο αιτιολογημένες γνώμες από ε, το Αυστριακό Κοινοβούλιο και από τη Γερουσία της Πολωνίας. Αυτά για σήμερα το πρωί. Θα συναντηθούμε εκ νέου στις 3 για μια μεικτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Κοντ και θα δούμε την ε, παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρακαλώ να είστε παρόντες, ε, επομένως να μην κάνουν την παρουσίαση και συνάδελφοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου με άδεια την αίθουσα.